Bene. Ε, Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω Ιταλικά, οπότε παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας. Να κηρύξουμε την έναρξη της ακρόασης αυτής της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτών. Και να καλωσορίσω τον υποψήφιο επίτροπο Τίμπορ Ναύρατσιτ να κάνω κάποιες αναρκτήριες παρατηρήσεις, διότι η ακρόαση αυτή, όπως θα ξέρει και εκείνο, είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική. Όχι μόνο όμως για την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω, αλλά και για την παρουσία των συναδέλφων από τις Επιτροπές Ήτρε και την Επιτροπή ΠΕΤΗ. Η Ήτρε είναι επιτροπή που θα συμμετάσχει, ενώ η Επιτροπή ΠΕΤΗ είναι απλώς παρατηρήτρια. Αυτός ο συνολικός, ο ομαδικός χαρακτήρας της ακροασίας μας δείχνει ότι ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα έχουν αξία αυταπόδεικτη ως αυτούσιες αρχές, αλλά και οικονομικές προεκτάσεις, καθώς και κοινωνικές. Έτσι λοιπόν οι εκπαιδευτικές πολιτικές και οι πολιτικές μάθησης έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες που θα προσφέρουμε στους νέους. Το ίδιο και για την πολιτική για τους νέους που είναι κεντρική σημασία για τη στρατηγική 2020. Αυτό σημαίνει ότι για μας τα θέματα αυτά είναι ζωτική σημασίας για την υλοποίηση των αρχών της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για να κατανοήσουμε ποιο είναι το όραμα της Ευρώπης που έχουμε σήμερα και ποιο ανθρώπινο, πολιτικό και κοινωνικό κεφάλαιο προτείνουμε στους πολίτες σήμερα. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Ναύρατσιτ, δεν πρέπει να υποτιμηθούν οι ανησυχίες, οι εκκλήσεις που μας έχουν απευθυνθεί τις τελευταίες ημέρες αλλά και αυτούς τους μήνες από πολλούς πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών. Σήμερα θα έχετε κάθε ευκαιρία και θα το φροντίσουμε εμείς αυτό σε αυτήν την ακρόαση να υπάρχει ο μέγιστος δυνατός αμοιβαίος σεβασμός. Θα έχετε λοιπόν κάθε ευκαιρία και το εύχομαι να μας καθησυχάσετε για το ότι και εσείς ε, ε, σέβεστε απολύτως τις αρχές της συνθήκης και ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές μας θα ε, χαραχθούν μέσα στην πλήρη ανεξαρτησία την προσωπική σας και στο ρόλο σας ως Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω Τη διαδικασία προβλέπεται σήμερα για την διεξαγωγή αυτή τη ακρόαση. Όπω τα γνωρίζετε, οι κατευθυντήρε γραμμέ για τι ακροάσει των υποψήφιων επιτρόπων περιλαμβάνονται στο παράδειγμα 16 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου, όπου λέγεται το εξή. Το Κοινοβούλιο αξιολογεί του υποψηφίου επιτρόπου βάσει των γενικών του ικανοτήτων, τη ευρωπαϊκή του δέσμευση και τη προσωπική του ανεξαρτησία αποτιμά τη γνώση του μελλοντικού χαρτοφυλακίου που θα αναλάβουν και τις δυνατότητες επικοινωνίας τους. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για την ακρόασή μας. Ε, σας ευχαριστώ κύριε υποψήφια Επίτροπε που ήδη απαντήσατε σε κάποιες προκαταρκτικές ερωτήσεις που σας απεστάλησαν. Οι απαντήσεις σας έχουν διανεμηθεί σε όλα τα μέλη, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Και συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο μετέγραφα για τη σημερινή ακρόαση μαζί με το βιογραφικό σας. Σε αυτό το σημείο θα έλεγα να οργανώσουμε τη συζήτηση ως εξής. Αρχικά, ο υποψήφιος επίτροπος Ναύρατσιτ θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει 15 λεπτά για τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις. Στη συνέχεια, όπως γνωρίζετε, θα έχει θα υπάρξει χρόνος για 45 ερωτήσεις από τους ε, συναδέλφους βουλευτές και η συζήτηση θα βασιστεί στην αρχή ping-pong όπως ονομάστηκε, δηλαδή παρεμβάσεις τριών λεπτών συνολικά η κάθε μια. Ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση του Επιτρόπου σε κάθε ερώτηση. Να θυμίσω ότι ο πρώτος γύρος ερωτήσεων θα τεθεί από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και από τους μη εγγεγραμμένους. Και ε, θα ακολουθήσει η Επιτροπή ΙΤΡΕ, η οποία συμμετέχει στην ακρόαση αυτή, ενώ η Επιτροπή Αναφορών πέτει είναι απλώς προσκεκλημένη. Μόλις ολοκληρωθεί ο γύρος ερωταπαντήσεων, στο τέλος ο υποψήφιος επίτροπος θα έχει πέντε λεπτά στη διάθεσή του για μια καταληκτήρια παρέμβαση και οι γλώσσες που θα καλυφθούν σήμερα από, την από τη Διερμηνία είναι 23. Μπορούν οι ομιλητές να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα τους εκτός από τα μαλτέζικα. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους. Η ακρόαση θα μεταδοθεί απευθείας στο διαδίκτυο του Κοινοβουλίου και επίσης εκεί θα υπάρχει και βιντεοσκοπημένη η ακρόαση. Επειδή θα μεταφράζεστε ταυτοχρόνως από τους διερμηνείς, παρακαλώ να μιλάτε με έναν φυσιολογικό ρυθμό. Να καλωσορίσω λοιπόν και πάλι τον κύριο Ναύρατσιτς και του δίνω το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Αγαπητοί Πρόεδρε, κυρία Κώστα, κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη του, είστε αυτοί που διαμορφώνετε τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν σας παρουσιάσω το δικό μου όραμα για αυτό το χαρτοφυλάκιο, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το λόγο που είμαι ευτυχής να βρίσκομαι εδώ απόψε. Το να είναι κανείς επίτροπος σημαίνει να είναι στρατευμένος Ευρωπαίος. Το να είναι κανείς επίτροπος σημαίνει να εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και κανένα άλλο συμφέρον. Το να είναι κανείς επίτροπος σημαίνει να υπηρετεί τον Ευρωπαίο πολίτη. Δεν μπορώ να σκεφτώ μεγαλύτερη τιμή, επομένως από το να ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα. Γνωρίζετε κι εσείς, γνωρίζω κι εγώ, ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουγγαρίας ε, διήλθαν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Διαφωνήσαμε για συγκεκριμένα σημαντικά ζητήματα και εκφράσαμε τις αντιθέσεις μας ε, με έντονο τρόπο, με ηχηρό τρόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως, μια από τις μεγάλες αρετές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι μας δίνει το χώρο να ε, αντιπαραβάλλουμε τις διαφορές μας ε, και να λύσουμε τις διαφωνίες μας, αλλά με τρόπο ανοιχτό, δημοκρατικό και ειρηνικό να βρούμε μία λύση ε, στις διαφωνίες μας, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, μας κάνει πιο δυνατούς και σαν χώρες μεμονωμένα, αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Εν τέλει, μας ενώνουν οι ίδιες ευρωπαϊκές αξίες. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου, Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για αξίες ε, στις οποίες είμαι βαθύτατα και προσωπικά δεσμευμένος. Απόψε θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το όραμα που έχω για την παιδεία, τον πολιτισμό, την νεολαία και την ηθαγένεια. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το έργο το οποίο πρέπει από κοινού να φέρουμε σε πέρας. Αν διαβάσετε ορισμένες από τις εφημερίδες μας, ίσως αποκομίσετε την εντύπωση ότι το εν λόγω χαρτοφυλάκιο δεν είναι και το πλέον επίγον. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ. Διότι ποια πρόκληση είναι πιο επίγουσα από το μέλλον της νεολαίας μας. Ποιο πρόβλημα είναι πιο ανησυχητικό από την ανεργία των νέων που παραμένει πάνω από το 50% σε ορισμένες χώρες. Ποιο καθήκον είναι πιο σημαντικό και πιο απαραίτητο από το να δώσουμε στις μελλοντικέ γενιές την καλύτερη δυνατή εκκίνηση ε, στη ζωή τους και τι μπορεί να είναι πιο πολύτιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την παιδεία, τον πολιτισμό της και την αίσθηση της ταυτότητας. Ποιοι τομείς πρέπει να τύχουν προστασίας ε, περισσότερο από τις πολιτισμικές διουρικές βιομηχανίες. Τι είναι η Ευρώπη αν δεν είναι κοινή κληρονομιά, μια κοινότητα κοινών αξιών. Αξιότιμοι βουλευτές, πιστεύω ότι το χαρτοφυλάκιό μας είναι όσο ζωτικό όσο οποιοδήποτε άλλο. Αν θέλουμε να επανοικοδομήσουμε μια δίκαιη βιώσιμη οικονομία πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση, με την παιδεία. Πρέπει να προετοιμάσουμε τους νέους μας για έναν πολυπολιτισμικό και ταχύως μεταβαλλόμενο κόσμο. Αν θέλουμε οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί μας να βρουν νέο ακροατήριο ε, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να τους δώσουμε τα εργαλεία για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να ανθίσουν στην ψηφιακή εποχή. Όλοι ε, θεωρούμε ότι η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η συμμετοχή στα κοινά είναι μέσω να απελευθερώσουμε το δυναμικό μας ως ανθρώπινα όντα. Δεν είμαστε οικονομικοί πόροι, δεν είμαστε εξαρτήματα σε ένα μηχάνημα. Είμαστε άνθρωποι, ανθρώπινα όντα, επομένω βρίσκουμε νόημα στις σχέσεις μας με τον πλησίον. Γινόμαστε ολόκληροι, ε, μια ολότητα, όταν συμβάλλουμε σε κάτι που μας υπερβαίνει, σε κάτι που μας ξεπερνά. Οι πολιτικές στο χαρτοφυλάκιό μας ε, υλοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, άρα στο δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες και έτσι πρέπει να είναι. Όμως συμφωνώ με όσους από εσάς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο. Πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκομένους φορείς να αντιμετωπίσουν τις επίγουσες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι. Θέλω λοιπόν να εξυγχρονίσουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα από ε, την ε, πρώην σχολική εκπαίδευση μέχρι τις μεταπτυχιακές σπουδές. Να έχουμε ε, άτομα ε, και δασκάλους ε, με σωστή κατάρτιση, με κίνητρα που να αναγνωρίζεται η αξία τους. Θέλω τα σχολεία, τα πανεπιστήμια να μάθουν τις νέες τεχνολογίες και να υιοθετήσουν νέους τρόπους διδασκαλίας και εκμάθησης και θα πρέπει να εκπληρώσουμε τους στόχους μας στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020, όλο και περισσότερους ε, αποφύτους ανώτερης ανώτατης εκπαίδευσης, ε, λιγότερη σχολική εγκατάλειψη, γιατί ξέρουμε ότι κάποιος που αφήνει το σχολείο και δεν έχει δεξιότητες ε, θα έχει σημαντικότερα κοινωνικά μειονεκτήματα από τους υπολείπους. Ποιε είναι οι πρώτε μου προτεραιότητε για την επόμενη πενταετία. Πρώτον, πρέπει η εκπαίδευση να μπει στο επίκεντρο των σχεδίων της Ευρωπαϊκή Ένωση για ανάπτυξη και θέσεις εργασία. Έξω και ο Ζαν Κλοντ μου ζήτησε να στηρίξω ε, τη δέσμη επενδυτικών μέτρων που θα παρουσιάσει εντός τριών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του σήμερα. Δεσμεύομαι ενώπιον σας ότι θα ε, συνεχίσω και εγώ και θα, ε, αυτές τις προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου αυτού όχι μόνο τώρα στην αρχή της εντολή, αλλά κάθε χρόνο, όταν δηλαδή θα κάνει τις προτάσεις της, τις συστάσεις αναχώρα στα τα κράτη-μέλη κομισιών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας να επενδύσουν στους δασκάλους, στις νέες τεχνολογίες, στις νέες διδασκαλίες, να εξυγχρονίσουν τις διδακτικές μεθόδους και την διδακτέα ύλη. Ακόμη και όταν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διορθώσουν τα δημόσια οικονομικά τους, είναι ζωτική σημασία να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους στην παιδεία και την κατάρτιση. Δεύτερον, θέλω να εξασφαλίσω ότι οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες θα μπορέσουν να ανθίσουν στον ψηφιακό κόσμο. Η Ευρώπη έχει ηγετική θέση στο δημιουργικό περιεχόμενο και είναι κάτι που πρέπει να μα κάνει περήφανο. Σήμερα δεσμεύομαι ενώπιον σα ότι καμία εμπορική διαπραγμάτευση οπουδήποτε στον κόσμο δεν θα υπονομεύσει το ρόλο τη παιδεία και τη μεγάλη σημασία τη δημόσια ενίσχυση. Θα ήθελα να σα αναφέρω τα λόγια του Jean-Claude Δεν θα θυσιάσουμε την πολιτιστική ποικιλομορφία, πολυμορφία της Ευρώπης στο βωμό του ελεύθερου εμπορίου. Και εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του καθεστώτος περί δημιουργού θα προωθήσει και τους καλλιτέχνε μας, του δημιουργού μας, αλλά και την πολιτιστική πολυμορφία που είναι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Όλες οι ευρωπαϊκές δράσεις θα σέβονται την ε, μοναδική φύση της παιδείας μα. Αυτό το ζητάει και η συνθήκη. Τρίτον, θέλω τα πανεπιστήμια μα να γίνουν τα καλύτερα στον κόσμο. Πρόκειται από ιδιαίτερα πολύτιμα ιδρύματα για την Ευρώπη, καθότι είναι πυλώνες της κοινωνίας μας και ζωτική πηγή καινοτομία. Στην Κεντρική Ευρώπη πριν το 1989 ήταν οχυρά ελευθερίας, κρατούσαν ζωντανή την ελεύθερη σκέψη. Σήμερα πολλά από αυτά τα πανεπιστήμια πρέπει να ανοίξουν τις θύρες τους στον έξω κόσμο και να προσαρμοστούν στις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να βοηθήσει να εξυγχρονιστούν τα πανεπιστήμια μας και να οικοδομηθεί μια νέα σχέση αυτών με την ευρύτερη κοινωνία. Θέλω το τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή παιδεία, έρευνα και επιχειρήσεις, να γίνει μια πραγματική εταιρική σχέση. Θα συνεχίσουμε επενδύουμε στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το ΕΙΤ, και στις δράσεις μας μαρις Σκλοντόσφκα Κιουρί. Το ΕΙΤ είναι ήδη ένα ρηξικέλευθο πρόγραμμα που ήδη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε την καινοτομία και είμαι ευγνώμων προ το Κοινοβούλιο που το στηρίζει αυτό το Ίδρυμα, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο για να γίνει μια μεγαλύτερη επιτυχία και οι δραστηριότητε του να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα το βάλω στο επίκεντρο τη χάραξη πολιτική ε, στην Ευρώπη, γιατί μια καλή πολιτική χρειάζεται σωστή έρευνα, χρειάζεται ενδείξει, στοιχεία. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα ε, υπηρετεί όλου τους τομείς πολιτικής. Ε, είναι πραγματικά το μυαλό ε, στο κέντρο της σκέψης μας και θέλω όλοι να μπορέσουμε να αποφεληθούμε από αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, τέταρτη μου προτεραιότητα. Θα συνεργαστώ στενά με την ε, συνάδελφό μου Μαριάν Τίσεν, Επίτροπο για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, ώστε από κοινού να κάνουμε πάντο δυνατόν για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μόνο τμήμα της λύσης πολύ σκληρή δουλειά πρέπει να γίνει και από τα κράτη-μέλη. Όμως ε, θα στηρίξω στεναρά όσες προσπάθειες ε, γίνουν ε, για τη στόχευση, των, στοχεύοντας μάλλον με τους πόρους μου ακριβώς την επίτευξη αυτής, αυτού του σκοπού. Και πιστεύω ότι από κοινού μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Με τη δική σας στήριξη και συνεργαζόμενοι με τα κράτη-μέλη μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους να κάνουν τη μετάβαση προς το χώρο εργασίας. Και αυτό το θα το πετύχουμε με εξυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και συστημάτων κατάρτισης για να μπορούν να τα ανταποκριθούν απαιτήσει τη αγορά εργασία του 21ου αιώνα. Θα στηρίξουμε επίση την ε, εγγύηση για την νεολαία. Ε, θα χρηματοδοτήσουμε νέε εταιρικέ σχέσει μεταξύ πανεπιστημίων, ε, παιδευτικών σχολών, επιχειρήσεων. Θα βελτιώσουμε την ποιότητα των περιόδων άσκηση και μαθητεία και θα δώσουμε στου νέου ανθρώπου όλα τα ωφέλη και τη άτυπη μάθηση. Εκτό αίθουσα δηλαδή. Πέμπτη μου προτεραιότητα θέλω να φέρω και την νεολαία της Ευρώπης ε, ε, μέσα στον κόσμο της χάραξης πολιτικής. Η νεολαία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ε, προκλήσεις άνευ προηγουμένου. Η οικονομική κρίση και έχει οδηγήσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την ανεργία σε πολλές χώρες έχει επίσης ε, ε, δημιουργήσει και σημαντικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τη θέση των νέων ε, στην κοινωνία. Οι πολλοί νέοι σήμερα είναι καλύτερα ενημερωμένοι, συνδεδεμένοι επίσης τα έλεγα σε σχέση με προηγούμενες γενιές χάρη στα νέα κοινωνικά μέσα, αλλά δεν θέλουν πολλές φορές να αρθρώσουν ισχυρό πολιτικό λόγο για την διαμόρφωση της αυριανής κοινωνίας και αυτό θέλω να το αλλάξω. Ο διαρθρωμένος μας διάλογος με την νεολαία έχει αποδείξει την αξία του, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να φτάσουμε να μπορέσουμε να έχουμε επαφή και με λιγότερο ε, ευνοημένους ε, νέους. Θέλω λοιπόν να αναπτύξουμε νέες πλατφόρμες για να φτάσουμε σε ένα εκατομμύριο νέους ανθρώπους την επόμενη πενταετία. Αυτό θα σηματοδοτήσει μια πραγματική αλλαγή στη συμμετοχική δημοκρατία και μια πραγματική στήριξη στις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να φτάσει τους νέους. Έκτη προτεραιότητα θέλω να ε, δώσω μια νέα ε, ανανεωμένη έννοια ε, στον όρο Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Δεν είναι λέξεις αυτές οι δύο, Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, λέξη μια συνθήκη. Είναι κάτι παραπάνω από ένα κοινό διαβατήριο, η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Είναι κάτι περισσότερο από το συμπλήρωμα της εθνικής υπηκότητας. Θέλω η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια να είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το ζήσει, να το ανασάνει κατά κάποιο τρόπο. Κάτι το οποίο μας εμπλουτίζει την καθημερινή ζωή, κάτι που βοηθά να οικοδομήσουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα ταυτότητα η οποία θα μπορεί ε, να ε, συνάδει με όλες τις άλλες ε, μορφές και όλες τις άλλες πτυχές ε, της προσωπικότητάς μας. Το ε, χαρτοφυλάκιό μας είναι η καλύτερη δυνατή αφετηρία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός, όλα μας τα προγράμματα, όλες μας οι πολιτικές δημιουργούν την αίσθηση της ηθαγένειας, του ανήκειν. Η ε, Ευρώπη για τους πολίτες, το πρόγραμμά μας θα δώσει συνειδητοποίηση για την κοινή ιστορία, τις κοινέ αξίες, θα κάνει τον κόσμο να καταλάβει τι κάνει για αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις λέξεις αθλητισμός, πολυγλωσία δεν θα τις βρείτε βέβαια στο τίτλο του χαρτοφυλακίου, όμως ανήκουν στο χαρτοφυλάκι, ανήκουν στα καθήκοντά μου και είμαι υπερήφανο που έχω ευθύνη για αυτά τα δύο ζητήματα. Για πρώτη φορά στον κοινοτικό προπολογισμό ο ευρωπαϊκός αθλητισμός ε, για όλους έχει πλέον 300 εκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή του για να προστατεύσει τα δικαιώματα των νεαρών αθλητών και παιδιών, για να καταπολεμήσει τη βία, τις διακρίσεις, το ντόπινγκ ε, και τα στημένα παιχνίδια. Θέλω να βοηθήσω το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας να δημιουργήσουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού και μπορείτε να βασίζεστε στην πλήρη μου υποστήριξη όταν θα δρομολογήσουμε του χρόνου την πρώτη τέτοια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Επίσης θέλω να σας πω και είμαι περήφανος γι' αυτό έχουμε ισχυρά εργαλεία για να προωθήσουμε την εκμάθηση γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία. Έχουμε το Erasmus Plus, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ένα από του βασικού έξι στόχου που έχει είναι η εκμάθηση γλωσσών, η γλωσσική πολυμορφία. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε, να αξιοποιήσουμε πλήρω τη μεγάλη αυτή ευκαιρία που έχουμε για να προωθήσουμε όλε τι γλώσσε τη Ευρώπη ανεξαρτήτω του αριθμού ε, των ανθρώπων που τι μιλούν. Ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων μα καλεί να σεβαστούμε τη γλωσσική μα ε, πολυμορφία και θα συνεργαστώ στενά με τον κύριο Τίμερμαν, ώστε πραγματικά να δικαιώσουμε τι φιλοδοξίε αυτού του χάρτη. Αξιότιμοι βουλευτέ ε, έχω μπροστά μου πολύ σημαντικέ προκλήσει και για να ανταποκριθώ σε αυτές θα χρειαστώ τη δική σας υποστήριξη. Ακόμη και αν επιτύχουμε, δεν θα δούμε σήμερα όλα τα ωφέλη, όπως οι αρχιτέκτες των μισιονικών καθεδρικών ναών μπορεί ίσω να μην ε, ζήσουμε για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα της δουλειά μας. Όμως είμαι έτοιμος για αυτό το χρέος που έχω να επιτελέσω και με, ε, ελπίζω να έλθετε κι εσείς μαζί μου σε αυτό το, το μονοπάτι. Ε, έτσι με μια νότα πιο αισιόδοξη. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να ενθαρρυνθούμε και να αντλήσουμε δύναμη από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα. Το Εράσμου είναι ε, εμβληματική εφεύρεση Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβολίζει σημαντικέ αξίε τη Ευρώπη, το ανοιχτό πνεύμα, την κινητικότητα, την επιθυμία να συναντηθούμε, να κατανοήσουμε των πλησίων μα. Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα μα βοηθάει το Εράσμου ε, να χτίσουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, κάτι που χρειάζεται η Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα φροντίσω και εγώ να τύχει της χρηματοδότησης που του πρέπει, ε, γιατί γνωρίζετε και εσείς και εγώ ότι ε, δεν είμαστε εμείς ε, οι δύο δηλαδή θεσμοί, τα δύο θεσμικά όργανα που διακινδυνεύουμε τη χρηματοδότησή του. Πρέπει λοιπόν, ε, γιατί ξεκινήσαμε νωρίτερα και το νέο πρόγραμμα, να φροντίσουμε ότι θα φέρει αποτελέσματα για τα 4 εκατομμύρια ανθρώπων που θα σπουδάσουν, θα εργαστούν ή θα δηλώσουν εθελοντέ σε μια ξένη χώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτέ είναι οι προτεραιότητέ με τα επόμενα πέντε χρόνια. Έχουμε πολλά να κάνουμε, έχουμε την άκρη να ακούσουμε του πολίτε. Θα είναι τιμή μου να εργαστώ για την ευρωπαϊκή υπόθεση, να υπηρετήσω την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, ω Ευρωπαϊκό Επίτροπο, ο Επίτροπο ο δικό σα. Α αρχίσουμε τη δουλειά σα. Ευχαριστώ.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 δεν συμμερίζεται τις ε, φιλελεύθερες αξίες της Ευρώπης. Με ποια μέτρα ε, προερχόμενος ε, από μια τέτοια κυβέρνηση σκοπεύετε να προωθήσετε την πολιτική ποικιλομορφία στην Ευρώπη και να στηρίξετε ακριβώς τον κλάδο αυτό και τους καλλιτέχνες. Thank you very much for the Ευχαριστώ για την ερώτηση. Εάν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 Εάν υπάρχουν τάσεις αντιευρωπαϊκές στην Ουγγρική εκπαιδευτική πολιτική, βεβαίως θα τις καταπολεμήσω ως, ως επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνάδελφος Κούρτσιο Μαλτέζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ναύρατσιτ, μιλάτε ως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 προσωπικός ανέκαθεν είχα πολύ καλές σχέσεις με τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ουγγαρία. Έχω εργαστεί για μη κυβερνητικές οργανώσεις και ως υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Δίκησης έχω δημιουργήσει μια ομάδα εργασία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, όπου συμμετέχουν και εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλη μια ομάδα εργασίας για την δικαιοσύνη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 πιστεύω στις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μεταξύ των οποίων είναι και ο πλουραλισμός στα ΜΜΕ. Και βεβαίω ε, ό,τι προβλήματα προέκυψαν τα τακτοποιήσαμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τροποποιήσαμε τον νόμο όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Εγώ ήμουν ο διαμεσολαβητής, εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις, κατέληξα σε συνένεση με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς γιατί προσωπικά πιστεύω στον πλουραλισμό στα ΜΜΕ. Ως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης νομίζω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 Κύριε Επίτροπε, εξ του ΕΛΚ ήθελα να πω ότι εκτιμούμε γεγονός ότι παρατηθήκατε από τη θέση του Υπουργού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 η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει όντως να αντιμετωπιστεί με τρόπο ενίο, όχι καταγερματισμένο, γιατί πρόκειται για ένα μόνο σύστημα που ξεκινά από τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό για να φτάσει στο πανεπιστήμιο και στα μετά το διδακτορικό διπλώματα.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 ή κάποιοι ήταν αντίθετοι μια εποχή. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ε, στην χώρα μου. Σε ό,τι αφορά αυτό το νόμο για τα μίντια, εγώ ήμουν διαπραγματευτής, ο οποίος τελικά κατάφερε την επίτευξη συμφωνίας. Και τροποποιήθηκε ο νόμος, ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Ε, Ευχαριστούμε ο συνάδελφος κ. Λέρος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 Να πω λοιπόν ότι μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών με διαπραγματεύσει τα πάντα μπορούν να βρουν τη λύση του. Ευχαριστούμε και τώρα η συνάδελφο Εύαν. Ευχαριστώ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 θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμε δεξιότητες ε, που θα προσφέρουν και ανταγωνιστικότητα. Και από την άλλη βεβαίω, υπάρχει και η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα ζητήσω την στήριξη του κυρίου Τίμπερμαν, του πρώτου αντιπροέδρου της Κομισιόν και θα καταγράψουμε την κατάσταση και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατεύσουμε τι μειονοτικέ γλώσσε.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 και τι συνηθισμένε πολιτικέ περικοπών σε όλα τα κεφάλαια του προπολογισμού και στη συνεργασία μας με τον μελλοντικό επίτροπο Ντομπρόφσκη. Τι ε, προτάσει θα υποβάλλετε ώστε να υπάρξει ενσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και εν ώψη της επίτευξης των στόχων της Στρατηγική Ευρώπη 2020 στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση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 στην χώρα σας ε, αντισημίτες συγγραφείς όπως ο Άλβερτ Βος, ο Ιωζεφ Νιερέ, Τσετσίλε Τομάη κλπ. είναι στη διδακτέα ύλη των σχολείων. 21% των Ούγγρων ε, συμπαθούν την είναι υπέρ της άκρας δεξιάς. Εάν γίνεται επίτροπος πολιτισμού, εκπαιδευση και νεολαία, τι να περιμένουμε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 ε, προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τι σκοπεύετε να κάνετε, έχετε συγκεκριμένε προτάσει για πραγματικέ επενδύσει στου παραδοσιακού πολιτισμού και ειδικά στον δημιουργικό τομέα. Σα ευχαριστώ. Ε, Νομίζω πως ε, το πρόγραμμα Erasmus Plus και η χάρτα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 με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης και δεδομένης, όπως είπα, και της οικογενειακής μου καταγωγής ε, έχω προσωπική αντίληψη για το θέμα και βεβαίως ε, θα επιμείνω σε αυτό το θέμα και θα προσπαθήσω να προωθήσω αυτές τις γλώσσες.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 Ένα από τα τους πιο σημαντικού τομεί όταν μιλάμε για την βελτίωση της mm. ανταγωνιστικότητας είναι πως ε, οι κοινότητες ε, γνώσης και καινοτομίας που διαμορφώθηκαν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 Κύριε Υποψηφί επίτροπε, θα ήθελα εγώ να αναφερθώ στην εκπαίδευση των αναπήρων παιδιών. Μιλάμε παντού για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 Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οι συστάσεις ε, των συνηγόρων του πολίτη να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και αυτό πρέπει να είναι και έργο και καθήκον της κυβέρνησης. Οι συστάσεις λοιπόν ε, του διαμεσολαβητή πώς θα εφαρμοστούν ε, και στον κανονισμό και στις διαδικασίες της Κομισιόν αλλά και σε όλα τα θεσμικά όργανα μεταξύ αυτών και στους εκτελεστικούς οργανισμούς. Ευχαριστώ. Δύο πράγματα θα αναφέρω από τη συνθήκη.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 την κάνετε μια από τους πρώτους στόχους σας και, την άμεση και, την, ε, και τις πρώτες σας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 και οι πρωτοβουλίε που θα αναλάβουν οι πολίτε να εξετάζονται πραγματικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να καταλήγουν και σε νομοθετικέ πρωτοβουλίε και κάποια χειροπιαστά τελικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών είναι ένα μέσο πολύ σημαντικό και προοδευτικό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 εκφέρει μπορεί, έχει τα μέσα. Και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Αν ένα μεμονωμένο άτομο, ή μια κοινότητα στην Ευρώπη θεωρεί ότι παρα... έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του ή της, υπάρχουν στη διάθεσή τους μέσα για να επανορθώσουν την κατάσταση.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 ευρωπαϊκά θεσμικά ιδρύματα. Οι πολίτε είναι πιο κοντά στι εθνικές δημοκρατίες που έχουν ιστορία εκατοντάδων ετών. Εδώ λοιπόν δεν φτάνει η νομοθεσία. Απαιτούνται επαφέ μεταξύ των ανθρώπων. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι το θεμέλιο της κοινή μα δημοκρατίας στο μέλλον. Η Επιτροπή σας λοιπόν θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει τα 28 έθνη της Ευρώπης. Αυτό εννοείται. Ναι. Mit említettem már korábban is. Όπως προείπα, κατά την άποψή μου, μία από τις βασικές αρχές, ένα από τα βασικά στοιχεία της όλης μου, ε, της όλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη είναι ε, το ενωμένη στην πολυμορφία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 για όλου του ευρωβουλευτέ από ποια γωνιά τη Ευρώπη και αν προέρχονται. Σε αυτό το σημαντικό στοιχείο πρέπει να επιμείνουμε. Και τώρα ο λόγο στην συνάδελφο Βίξτρομ από την Επιτροπή Αναφορών. ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ναύρατσιτς, δεν είμαι εντελώ ικανοποιημένη, ούτε επίστηκα πλήρω ε, από τι απαντήσει που έχετε δώσει μέχρι τώρα στου συναδέλφου μα, επειδή την τελευταία δεκαετία έχετε ε, υπάρξει ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της σημερινής Ουγγρικής Διοίκησης ε, ως ε, αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας και ως υπουργός της κυβέρνησης Φίντες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 πολιτική. Θα ενθαρρύνεται μήπως τις ΜΚΟ για να ενισχύσουν ακριβώς ε, την ε, ευρωπαϊκή υπηκότητα. Κοιτάξτε, προσωπικά, εγώ ήμουν ε, και υπέρ των ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά ξεκινήσαμε και ένα πρόγραμμα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 να βρεθεί η πολυγλωσία είναι σημαντικό δικαίωμα, θεμελιώδη δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλέ φορέ ε, το επικαλούνται και οι αναφέρονται στην Επιτροπεριφερειών ω πρόβλημα. Δυστυχώ όμω ε, είναι πολλά τα κενά και τα προβλήματα. Παραδείγματο χάρη, ε, έχουμε τρει γλώσσε εργασία, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, στα δικαστήρια και ιδίω ό,τι αφορά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 συναλλαγές που έχουν ε, με το κράτος. Μιλάμε δηλαδή για κάποιου κρατικούς φορεί, θα πάντων επίσημου φορεί, στους οποίου μπορούν να στραφούν οι άνθρωποι αυτοί και να μπορούν να μιλήσουν τη μητρική τους γλώσσα. Υποψήφιε επίτροπε στο πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες ε, έχουν ε,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 και υπό την ιδιότητά του ως μέλους της Επιτροπής Ήτρε, την κυρία Κριστίνα Λιμπάτσκα. Ε, ε, Κύριε υποψήφιε επίτροπε, μας ε, διαβεβαιώσατε επανειλημμένως πως ε, παρατηρήσετε τις εξής Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα όσα αναφέρονται στις συνθήκες. Και όμως ε, προσφάτως ο κύριος Όρμπαν είπε το εξής. Επιλέξει. Θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε νέες σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησής μας και του Ούγκρου Επιτρόπου και αναμένω πως ο Ουγγρος Επίτροπος θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας στις Βρυξέλλες. Κλείνουν τα εισαγωγικά.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 για τα συμπεράσματά σας ε, πριν, ε, λήξουμε, πριν κηρύξουμε τη λήξη της ακρόασης. Ευχαριστώ λιγότερο από πέντε λεπτά. Κυρία Κώστα, ε, αγαπητέ, και αγαπητοί βουλευτέ. Σα ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσω το δικό μου, τη δική μου θεώρηση αυτού του χαρτοφυλακίου. Ελπίζω ότι υπήρξα σαφή για τι προτεραιότητέ μου για την ερχόμενη πενταετία. Απόψε είχαμε μια ειλικρινή και ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων. Έτσι θα πρέπει να γίνεται πάντοτε. Αυτό είναι η δημοκρατία στην πράξη. Και έτσι θέλω να είναι και η σχέση μα και έτσι να εξακολουθήσει. Από την αρχή της ακρόασης δήλωσα ότι είναι τιμή μου να εξυπηρετήσω τον ευρωπαϊκό ε, σκοπό και αυτήν την ε, επιτροπή. Τρεις ε, ώρες αργότερα και 45 ερωτήσεις αργότερα δεν άλλαξα γνώμη. Ίσα ίσα έχω πιστεί περισσότερο από πριν ότι μπορούμε να έχουμε μεγάλα επιτεύγματα και να επιτύχουμε μεγάλα πράγματα εφόσον συνεργαστούμε. Το κοινοβούλιο αυτό έχει συμβάλει σε μερικά από τα μεγαλύτερα στοιχεία της Ευρώπης σήμερα, από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες. Το Erasmus Sin το Creative Europe, τον πρώτο προπολογισμό για τον αθλητισμό. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν όλους σας για αυτήν την στήριξη, διότι κάποια από τα προγράμματα αυτά δεν, είχαν, δεν ήταν σίγουρο ότι θα έχουν έσει ο πέρας. Χάρη στη δική σας όμως τη συμβολή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορέσαμε να προβλέψουμε και τα ανάλογα κονδύλια για να υλοποιηθούν. Αν με εγκρίνετε λοιπόν ως Επίτροπο αυτό το πνεύμα συνεργασίας θα υλοποιηθεί από την πρώτη στιγμή της θητείας μου. Θα είναι προτεραιότητά μου ανα με την πρώτη ευκαιρία να επισκέπτομαι την Επιτροπή σας για να συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων το διάλογο που ξεκίνησε σήμερα. Ε, ελπίζω ότι ο διάλογος που θα έχουμε και στο μέλλον θα είναι εξίσου έντιμος και ειλικρινής όπως ήταν σήμερα. Σας ευχαριστώ. Allora, io desidero ringraziare και εγώ να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τις ερωτήσεις τους, τους συναδέλφους των Επιτροπών Κούλτ, Ήτρα και Πέτη, τον κύριο Ναύρατσιτς για τις απαντήσεις του και να πω ότι η ατμόσφαιρα που επικράτησε σε αυτή την ακρόαση νομίζω ότι ήταν αμοιβαίου σεβασμού με κάπως λίγο πιο ξεμένους τόνους κάποιες φορές, αλλά αυτό είναι και παιχνίδι του δημοκρατικού διαλόγου. Ήταν νομίζω ειλικρινής και ανοιχτός ο διάλογος που είχαμε και ε, καθόλου δεν προσπάθησε κάποιος να διαφύγει από τις απαντήσεις που του ζητήθηκαν. Θα ε, αποτιμήσουμε κάποια στιγμή την ακρόαση αυτή. Να θυμίσω λοιπόν στους συντενιστές και αντιπροέδρους ότι θα συναντηθούμε αύριο το πρωί σε ε, διακλεισμένο των θυρών συνεδρίαση για να αποτιμήσουμε αυτή την ακρόαση. Και αποχαιρετώντας σας να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μας της γραμματείας αλλά και τους διερμηνείς που τόσο πολύ κουράστηκαν και συνέβαλαν τα μάλα στην ακρόασή μας και προστατεύουν βεβαίως και την γλωσσική, ε, την γλωσσική πολυμορφία σε αυτό το κοινό.